Έχουν διανεμηθεί τα συνοπτικά πρακτικά. Αν δεν διαφωνεί κανεί, ε, εγκρίνονται και προχωρούμε στις ψηφοφορίες τώρα. Η πρώτη μας ψηφοφορία αφορά